Κοινοβούλιο. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι βάσει του άρθρου 74 του κανονισμού μαζί με τον Προεδρεύοντα του Κοινοβουλίου υπέγραψα τον κανονισμό για την ε, ε, μεταφορά για την κυκλοφορία οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών. Τα πρωτόκολλα, τα, τα πρακτικά